Καθίστε παρακαλώ για να αρχίσει και η συνεδρίαση. Our, uh, President, uh, ο πρόεδρος μας, ο Αλάν Λαμασούρ, έχει γονικά καθήκοντα σήμερα το απόγευμα. Ε, αδυνατή να παραστεί στην απογευματινή συνεδρίαση, ε, στην οποία κυρίως, ε, την οποία συγγνώμη, κυρίως θα αφιερώσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ, φροντίστε να έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, λάβετε θέσεις. Το πρώτο σημείο που είχε προβλεφθεί στην μέση διάταξη ήταν το 11, δηλαδή η κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το Κοινοβούλιο. Αποσύρθηκε αυτό, αναβλήθηκε. Στις 10 Απριλίου θα γίνει ψηφοφορία. Το συζητήσαμε στους συντονιστές ε, και τελικά κατέληξε ε, πρέπει να καταλήξει το Προεδρείο συμφωνία για την κατάσταση ακριβώς ε, των προβλέψεων ε, πρωτού γίνει ψηφοφορία. Προχωρούμε. Σημείο 12. Διαπραγματεύσεις για το Πουδοπού 2014-2020. Έκθεση, μάλλον αναφορά σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντιληφθούν και μελλοντικέ προοπτικέ. Ε, Συγητή Jean-Luc Ντεάνε και Ιβάιλο Κάλφιν. Ε, Ουδή είναι εδώ θα ε, με βοηθήσετε, ελπίζω να τα πω σωστά. 100 τροπολογίες κατατέθηκαν ε, από την Ήτρε και από την Επιτροπή Γυναικών και από την ΑΦΚΟ βάσει του άρθρου 50 ε, η Ρέτζι Λίπλ και Έμπλε, Λίμπε συγγνώμη, και Έμπλε ε, εξέδωσαν γνωμοδοτήσεις. 50 ήταν οι συμβαστικές που προετοίμασαν οι συνεισηγητές. Ας περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία λοιπόν. Ήθελα μόνο να εξηγήσω κάτι πρωτού αρχίσουμε. Ε, πρώτα θα ψηφίσουμε τις ε, συμβαστικές, ε, αντίθετα με αυτό που κάνουμε συνήθως, δηλαδή όταν, με τη σειρά όταν φτάνουμε σε αυτές διότι υπάρχουν διάφορες τροπολογίες επιτροπών που δεν είναι απαράδεκτες, οπότε δεν ε, πρέπει να σας ενημερώνω κάθε φορά. Θα είναι σχετικά ε, σύντομη η ψηφοφορία, εκτός και να ανακύψουν ε, κάποια προβλήματα που δεν νομίζω. Πρώτη συμβαστική των συνσηγητών είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 2 για την αιτιολογική D, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 για την πρώτη παράγραφο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 για την παράγραφο 2, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 για την παράγραφο 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 για την παράγραφο 4 Κατά τμήματα το ζήτησαν οι πράσινοι. Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει για την πρώτη συζήτηση, ε, ε, πρώτη αράδα, συγγνώμη, της συμβαστικής τροπολογίας. Ε, για την πρώτη πρόταση. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, ε, γκρίνεται. Ε, υπόλοιπη παράγραφος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. η συμβαστική 7 για την παράγραφο 5, υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 για την παράγραφο 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 για την παράγραφο 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9α, νέα παράγραφος, ε, για την παράγραφο 17α, νέα υπέρ παρακαλώ για τη συμβαστική 9α κατά αποχέ εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 10 για την παράγραφο 19 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 11 για την παράγραφο 20α και πάλι νέα παράγραφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12, παράγραφη 21 και 21α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η συμβαστική 13, παράγραφος 22, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 14, παράγραφος 23β νέα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Προχωρούμε. Στην πρώτη τροπολογία που πρέπει να ψηφίσουμε είναι μια προφορική τροπολογία των συνεισηγητών ε, που διαγράφει τον όρο strongly στην τροπολογία 42. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ, της προφορικής τροπολογίας υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η, η 43 αποσύρεται και άλλη μια προφορική τροπολογία για 44 των συνεισηγητών. Ε, αντί για στους συνομοθέτες λέμε νομοθετική αρχή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 45 το πρώτο τμήμα της 45 πρέπει να το ψηφίσουμε. Το δεύτερο καλύπτεται από συμβαστική 7. Υπέρ του πρώτου τμήματος ε, της τροπολογίας 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 59 Χέλγα είπε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι πράσινοι απορρίπτουν τη δική τους τροπολογία ακόμη και αυτή. Προχωρούμε στην προφορική τροπολογία για την τροπολογία 63 της κυρίας Γκρέσελ τι λέει η προφορική τροπολογία. Αντικαθιστά την τελευταία πρόταση και λέει διακρίνει την ανάγκη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να βασιστεί στην εκτιθή σε εμπειρία και να συμμετέλθει τον, ε, όλων των ε, ε, διαθέσιμων μέσων ώστε να σεβαστεί το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων ώστε να ληφθούν περισσότερο υπόψη απόψεις στο Κοινοβουλίο. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας, κατά συγκρίνεται. Η 63 ε, καλύπτεται ήδη από το άρθρο 4. Προχωρώ στην 65. Εδώ έχουμε προφορική τροπολογία πάλι από τους ε, συνεισηγητές. Λέει εκεί, είναι νέο το κείμενο, ε, ε, αυτό συνιστά σαφή αντίθεση προς τους συνθήκε και τι το του Κοινοβουλίου βάσει τη συναπόφαση και του δικαιώματο τροποποίησης ε, ισότιμα με το Συμβούλιο. Ε, έτσι λέει η τροπολογία υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 68 προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών Θέλει κάποιος από τους σοσιαλιστές να την παρουσιάσει. θα την διαβάσω εγώ απλώς. Ε, την προστίθεται στην παράγραφο 15 για την ε, γεωργική πολιτική και πολιτική συνοχής ε, υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται. Πάμε τότε στην 71 τρίπελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, η 72 πάλι της τρίπελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και πάλι ε, τώρα πάμε στην αύκο 7 μεικτή αρμοδιότητα υπέρ το άρθρο 7 κατά αποχές εγκρίθηκε Γιάν. Ε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν το είπατε, αλλά για την 87 ε, είχα καταθέσει προφορική τροπολογία. Ε, και εγώ δεν κρίνω ότι συμπεριλήφθηκε τελικά συμβαστική τροπολογία, παρότι μπορούσε να γίνει παραδεκτή και άρα την καταθέτω εκ νέου. Και βλέπετε το κείμενο στον κατάλογο στις ψηφοφορίες. Θέλω να υποβληθεί σε ψηφοφορία, παρακαλώ. Ε, πρόεδρος, ε, ολόκληρη, ακέραια την καταθέτεται. Είχα καταλάβει ένα τμήμα. Σα είπα ότι είναι στον κατάλογο ψηφοφορίας, αλλά έχω δικό μου κατάλογο ψηφοφορίας σε τροποποιημένο, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, στην αρχική 87 ε, είχα την ακόλουθη πρόταση. Ε, πιστεύει ακράδαντα ότι ο πενταετής ε, κύκλος του πολυδιετούς πλαισίου ενισχύει την νομιμότητα, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των δημοσιονομικών πόρων και αποτελεί προπόθεση για ενισχυμένο πολιτικό διάλογο. Αυτή είναι η αρχική μου πρόταση, δεν συμπεριλήφθηκε συμβαστική και θέλω να υπο Βάλω εκ νέου αυτή την τροπολογία όπως σας τη διάβαζα σε ψηφοφορία παρακαλώ. Ναι, ως προσθήκη μπορούμε να την ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 87 λοιπόν. Κατά. Νομίζω θα χρειαστεί ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ. 47 πρέπει να την ψηφίσουμε ως προσθήκη και μετά να ψηφίσουμε δηλαδή για το πρώτο τμήμα, για την πρώτο τμήμα της 87 λοιπόν παρακαλώ ε, να το αναφέρετε στο νέο κατάλογο ψηφοφορίας ε, και μετά ε, θα συνεχίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, πέρασε, εγκρίθηκε και τώρα για το σύνολο του κειμένου αφήνεται να καταπέσει, δεν το υποβάλλετε. Ναι, ναι, όντω, λέει ο κ. ε, μπορεί να καταπέσει το δεύτερο τμήμα, δεν ε, ε, επιμένω. Ωραία, 92 τότε. Έχουμε μια προφορική τροπολογία και λέει «Τονίζει την ανάγκη να τονώσει έναν ανοιχτό και ευρύ διάλογο για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσης και κυρίως την αποτίμηση αυτών. Παρακαλώ υπέρ». Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 ναι, των ε, συνσηγητών και πάλι Ε, που μεταπτωπίζει, αν καταλαβαίνω καλά, την ε, τροπολογία. Πρέπει να την ψηφίσουμε, έτσι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 94 γέραν φάρμ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95. Προφορική τροπολογία των συνεισηγητών και εδώ ε, προσθέτουμε το review. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 τώρα. Κλεις Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 97. Χέλγα Τρίπελ. Και 98. Α, αποσύρθηκαν και οι δύο. Είναι 98 και 97 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 μπέργκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές γκρίθηκε. Ωραία. Ε, Τιολογικές σκέψεις. Πρώτο, πρώτη, ε, πρώτη τροπολογία, Χέλγα Τρίπελ. Κατά τμήματα προτείνουν, ε, ε προτείνει ο εισηγητής. Τρία διαφορετικά τμήματα. Πρώτη τροπολογία, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δύο. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται ε, παλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Closed. Πέρας. Εγκρίθηκε. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα, το μεσαίο. Και το τρίτο και τελευταίο υπέρ. Κατά. 3. Κλέι υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 4. Τρίπελ υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 11. Τρίπελ υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 τρίπελ και πάλι είπε. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 15 ε, Μούλτερ Γένσεν υπέρ. Κατά. απόχέ. Ε, εγκρίνεται. Αύκο 1. μεικτή αρμοδιότητα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυκό και πάλι μεικτή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις νομοδοτήσεις. Εδώ θα κάνουμε μια αρχική οριζόντια ψηφοφορία ε, για το σύνολο των τροπολογιών που φέρουν επί των γνωμοδοτήσεων ε, που υπάγονται στο κυρίω πεδίο εφαρμογής ε, γιατί σχετίζονται με μονομένα προγράμματα και όχι με το ευρύ ζήτημα των διαπραγματεύσεων για το πολιετέ δημοσιονομικό. Ζητώ από τις ομάδε το εξή να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες που δεν εγγράφονται στο ε, κυρίως πλαίσιο της ε, γνωμοδότησης. Ζητώ από τις ομάδες να μου πούνε ποιοι είναι υπέρ του να ψηφίσουμε τις μεμονωμένες ψηφοφορίες και ποιοι, θα είναι, ε, και κατά. Με σαμποτάρετε, είστε κατά, απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, ο Σαλβαντόρ είναι κατά. Ε, τώρα, όσε τροπολογίε σχετίζονται με τα μεμονωμένα προγράμματα και όχι με το ευρύτερο πλαίσιο, ε, καταπίπτουν μετά από αυτήν την πρώτη ψηφοφορία και τώρα πάμε στην ΕΜΠΛ 2, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, ΕΜΠΛ 5, Πόνο το πρώτο και το τρίτο τμήμα θα ψηφίσουμε. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται και το τρίτο και τελευταίο υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Πάμε με βήμα ταχύ στην 20, 20 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Και τώρα Πάμε στην τελική τροπολογία λίμπε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία για την τροποποιημένη έκθεση με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται. Λείπει κάποιος. Μέχρι 31 πάμε. Πέρας. 25 είναι υπέρ. Εγκρίθηκε. Ε, ευχαριστώ που με βοηθήσατε και χάρη σε αυτό ε, ήταν ε, ομαλή η ψηφοφορία γιατί είχα ανησυχήσει πρέπει να το ομολογήσω. Πάμε τώρα στις μεταφορές των πιστώσεων. Uh, η συγκεκριμένη κυρία Γένσεν θέλει να πει κάτι για τη μεταφορά 660 εκατομμυρίων για, με τον 11031 για τα αλληλευτικά σκάφη. Θέλετε να πείτε κάτι. Νομίζω είναι σαφές υπάρχει η συμφωνία πλέον και πρέπει να μεταφερθούν τα κονδύλια για να ισχύσει και η συμφωνία όπως πρέπει. Οπότε είμαστε υπέρ. Ωραία λοιπόν, να ψηφίσουμε για τη μεταφορά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε και άλλη μια μεταφορά. Μεταφορά του Ευρωκοινοβουλίου. 65.000 ευρώ. Μόνικα, θες να πεις κάτι. Ευχαριστώ. 65.000 είναι. Αφορά ένα συνεργάτη του Κοινοβουλίου ε, που βγαίνει προώρα στη σύνταξη και μεταφέρεται το ποσό αυτό στην αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού για τους συνταξιοδοτούμενους υπαλλήλου. Να πω και για το δεύτερο μέσο τώρα, για την άλλη μεταφορά. Ωραία. Πρόκειται για το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο προτίθεται να κάνει μεταφορά πιστώσεων αντίστοιχη από την προμήθεια, αρχιοθέτηση και παραγωγή βγαίνει αυτό το κονδύλι και προστίθεται σε μία άλλη υποκατηγορία που είναι η ε, εμπειρογνώμονες για τον οικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό. Δεν είχε προβλεφθεί αυτή η δαπάνη στην αρχή, εξού και με τη φορά τώρα των πίστος; Okay. Right. So... Ωραία. Οπότε ψηφίζουμε για την μεταφορά για τις ε, συντάξεις των προπολογισμών του Κοινοβουλίου. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία. Κοινοποίηση προς την EBA. Μας το εξήγησε η Μόνικα. Πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό, Μόνικα. Με συγχωρείτε, ένα λάθος στην προηγούμενη ψηφοφορία. Το αίτημα προς το ελληνικό συνέδριο. Υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία. Υποβολή εκθέσεων για την αύξηση στο Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 71. Θέλετε να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, προσέξτε το είπα και στους συντονιστές την περασμένη εβδομάδα. Υπήρξε μια συζήτηση και μια συμφωνία επιτέλους με το Συμβούλιο. Όπως ξέρετε διαπραγματευόμαστε τώρα για να αυξηθεί το κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν στη διάθεσή τους ε, κονδύλια μέσω ενισχύσεων και εγγυήσεων για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να έχουν και μια ρευστότητα. Έχουμε μια μικρή διαφορά με το Συμβούλιο για το ε, τι θα γίνει με τα μερίσματα που μπορούν να προκύψουν από τη διαχείριση αυτών των ε, ε, ταμείων και των κονδυλίων. Επειδή δεν συμφωνήσαμε, προτιμήσαμε να τα αφήσουμε στην άκρη αυτό και να δούμε πότε θα πάρουμε την απόφαση αυτή σε προσεχές μέλλον, σε απότερο χρόνο. Και το αφήνουμε αυτό στην άκρη γιατί θα πρέπει κατεπηγόντως να εγκρίνουμε την έκθεση. Αλλιώς δεν θα προλάβει να πάει στην Ολομέλεια του Απριλίου και δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να μπλοκάρουμε το θέμα αυτό, ούτε το Συμβούλιο, ούτε το Κοινοβούλιο. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, για τις μικρομεσαίες και συμφωνήσαμε σε αυτό το συμβιβασμό να αφήσουμε το συγκεκριμένο θέμα στην άκρη, ε, αλλά να αποφασίσουμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μέσω ε, ενός δημοσιονομικού κανονισμού ή δεν ξέρω πώς αλλιώς, πώς ε, θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα το μέρισμα το συζήτησαν οι συντονιστές, συμφώνησαν καταρχήν, αλλά θα πρέπει και τυπικά τώρα να ψηφίσει η Ολομέλεια της Επιτροπής μας. Θέλει κανείς άλλος να σχολιάσει για την έκθεση της ΕΙΝΤΕ. Αλλιώς ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, 28 ψήφισαν. Πέρα τη ψηφοφορία. 26 υπέρ, 2 κατά. Έχουμε ακόμη ένα άλλο ζητηματάκι. Έχει να κάνει με την προφορική ερώτηση που συζητήθηκε το πρωί. Πάλι αν και η Θες να μας εξηγήσεις αν. μας αυτό το πρωινό. Ναι. Καλά, αυτό το θέμα γνωρίζετε ότι το έχουμε ξαναδεί στην Επιτροπή μας και το έχουμε ξανασυζητήσει. Όπως το, ε, ξέρετε, για τις πληρωμές, ιδιαίτερα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ε, λαμβάνουμε ειδοποιήσεις και στην εξωτερική πολιτική γενικά υπάρχει πρόβλημα πληρωμών παντού στον προπολογισμό και νομίζω στην περασμένη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ακούσαμε τους αρμοδίους επιτρόπους προεπολογισμού και αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά θεωρήσαμε ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει στην Ολομέλεια δημόσια συζήτηση και να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα από, την, από ότι σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Στην τελευταία συζήτηση, στην τελευταία Ολομέλεια της χρονιάς για μας, να δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και ιδιαίτερα στον τίτλο 4 και στην ανθρωπιστική βοήθεια βοήθεια. Να δημοσιοποιηθεί περισσότερο αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό προτείνουμε να γίνει προφορική ερώτηση με συζήτηση στην Ολομέλεια. Και αυτό που πρέπει τώρα είναι να το εγκρίνουμε. Okay. Ωραία. Γιώργη, ναι, να πω απλώ ότι στη συνάντηση, των συντονιστών Τη συζητήσαμε την ερώτηση αυτή και είπαμε ότι η αναφορά στο CFSP δεν θα πρέπει να υπάρχει, αλλά να αναφερθούμε στην Ουκρανία, στην κατάσταση της Ουκρανίας και για τη στήριξη του πακέτου προς την Ουκρανία. Κύριος Χάρτοχ, θα ήθελα να πω ότι αυτό ε, τίθεται ως ερώτημα εξ ονόματος της Επιτροπής Προπολογισμών, αλλά βγάλετε το δικό μου όνομα, δεν είναι εξ ε, του βουλευτού κυρίου Χάρτον. Okay, your, request is Εντάξει, το σημειώνουμε και θα το λάβουμε υπόψη. Απλώς να ξεκαθαρίσουμε. Για την Ουκρανία το συμφώνησαν οι συντονιστές όσων Κατάλαβα, ναι. Αλλά νομίζω ότι ήταν ε, αποδεκτό να γίνει αυτή η μνήμα. Ωραία. Να ψηφίσουμε τότε. Είναι ερώτηση της Επιτροπής με την εξαίρεση του συναδέλφου από την Ευρώπη της Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Όχι, ωραία, με τα χειρών. Υπέρ της προφορικής ερώτησης. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία. Συνεχίζουμε με τα κτίρια. Χρειάζεται να ψηφίσουμε εδώ. Μόνικα. Θέλεις να μας ενημερώσεις. Να μας πεις ε, τι θα γίνει και πώς ε, θα ψηφίσουμε. Έχω να πω μερικά πράγματα όντως. Λοιπόν, το πρώτο, πολύ προσφυλές μας θέμα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής σε αντίθεση με την περασμένη πρόταση η τωρινή είναι καλή και ε, αποδεκτή και η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και η ίδια η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να βρούνε κάποιους λογικούς όρους παρά την πόλη του Λονδίνου ε, για να μην ε, ξεσπάσουμε σε λιγμούς μόλις δούμε τα αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε ένα νέο κτίριο τώρα για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή γιατί για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της και υπόσταση καν χρειάζεται δικό της κτίριο η ΕΜΠΑ. Οπότε ε, πρόκειται για το κτίριο Canada Square 1 το οποίο έχει μισθωθεί 4.153 τετραγωνικά τα μισά είναι ε, γραφεία 12 της διάρκεια της μίσθωσης και στο ίμιση της περίοδου υπάρχει η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης με 9 μήνες ε, προθεσμία. Από το 14 μέχρι το 26 λοιπόν είναι αυτό το διάστημα και τον άλλο μήνα, τον Απρίλιο, θέλουν να έχουν υπογράψει όλα τα δικαιολογητικά και τα μισθωτήρα συμβόλαια για να αρχίσει η λειτουργία το Μάιο. Πρόκειται να μεγαλώσει και σε μέγεθος η ΕΜΠΑ. Βέβαια ακούμε διάφορα στοιχεία διαφορετικά ε, ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεγαλύτερα η ΕΜΠΑ, αλλά ακόμα και αν δεχτούμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το εμβαδόν δεν είναι υπερβολικά μεγάλο, είναι λιγότερα ε, οι χώροι γραφείων που αναλογούν στους εργαζομένους σε σχέση με τους εργαζομένους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 31 τετραγωνικά αναλογούν σε κάθε εργαζόμενο και 35 συνολικά εκτός από το γραφείο του, τουαλέτες, κοινόχρηστη χώρη κτλ. Το κόστος πώς είναι. Ε, ετήσιο μίσθωμα 2,18 ε, εκατομμύρια, αλλά έχουμε 32 μήνες χωρίς υποχρέωση καταβολής ενοικίου. Δηλαδή 5,676 εκατομμύρια ουσιαστικά μας χαρίζουν για αυτή τη 12 ετία και ανά τετραγωνικό αν το υπολογίσουμε είναι 398 ευρώ άδειο και 503 με τον εξοπλισμό και με τα διάφορα έργα και με διάφορα μικροέξοδα και δαπάνες που χρειάζονται πάντα για κατασκευές. Πάντως ε, είναι κάτω από 600 ευρώ ε, που για το Λονδίνο που είναι ακριβή πόλη νομίζω ότι είναι ένα λογικό ποσό. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι <laughs> πανάκριβο το Λονδίνο και ε, πραγματικά αυτό το κτίριο κοντά στο αεροδρόμιο είναι ένα καλό, σε καλή κατάσταση, όχι πολυτελές, αλλά είναι εντάξει, προσφέρεται και από λειτουργικότητα και από ε, περιβαλλοντικές μελέτες, έχει πολύ καλές επιδόσεις και επιτρέπει και ευελιξία αν χρειάζεται επέκταση ή και μείωση των χώρων υπάρχει αυτή η ευελιξία. Κάτι και το μοναδικό που έχω εγώ να επικρίνω είναι το CBRE, οι σύμβολοι αυτοί που λέγουν ότι είναι 570.000 το κόστος για τους συμβούλους. Να το προσέξει παρακαλώ αυτό και η Κομισιόν και η ΕΜΠΑ. Ε, να μην πληρώνουμε δικηγόρους και συμβούλους ε, τόσο ακριβά. Υπάρχει μια πρακτική στις τράπεζες που είναι πολύ χαμηλότερο το κόστος. 570.000 ευρώ για νομική συνδρομή συν 53.000 δεν ξέρω Κάποιοι άλλοι δικηγόροι, 600.000 είναι πολλά τα λεφτά. Και αυτό είναι για μένα το απαράδεκτο. Και το, ε, θέλω να το δηλώσω να γραφεί και στα πρακτικά. Μην το δούμε πουθενά μπροστά μας. Πάνω από 600.000 δίνουμε για νομική συνδρομή και για παροχή συμβουλών. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Κατά τα άλλα, ε, είναι το κόστος αρκετά συμμαζεμένο. Το προβληματικό κεφάλαιο ποιο είναι. Την περασμένη φορά είχαμε κάνει κάποιες γραπτές παρατηρήσεις για το σύμβολο αυτό το CBRE ε, και το έχουμε κατονομάσει στην προηγούμενη μας ε, απόφαση, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Από πλευράς μου λοιπόν θα μπορούσα τώρα να δώσω το ok για το κτίριο αυτό, γιατί πραγματικά είναι σε λογικά πλαίσια, είναι ένα κτίριο που μας βολεύει και γενικά έχει ένα συμμαζεμένο κόστος το οποίο μπορούμε και προς τα έξω να υπερασπίσω. I have... Uh, Εντάξει. Έχουμε και ακόμη κάποιους συναδέλφους. Η κυρία Τσορμποπαχάτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είχαμε προβλήματα στο παρελθόν με αυτό το οργανισμό. Η ερώτηση είναι Σίγουρα, αν είμαστε συστηματικοί και υπομονετικοί, θα μπορέσουμε να πείσουμε τους οργανισμούς να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που διαθέτουν αποτελεσματικά. Χαίρομαι λοιπόν που αφιερώσαμε χρόνο και προσπάθεια σε, αυτήν την, σε αυτό το εγχείρημα. Είχε αποτέλεσμα και ελπίζω ότι και άλλοι θα διδαχθούν από αυτήν την εμπειρία. Δεν θα προσπαθούν να παρακάμπτουν την Επιτροπή Προπολογισμών για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ γιατί υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από αυτή την πρόταση. Ωραία λοιπόν. Θα ψηφίσουμε να μην υπάρξει νομοδότηση από αυτού. Σωστά. Οι συνάδελφοι λοιπόν ας ψηφίσουν υπέρ του να μην έχουμε νομοδότηση. Όσοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ωραία, νομίζω ότι εγκρίνεται. Και για το σπίτι της Ευρώπης υπάρχει κάτι ακόμη. Ναι, πρέπει να μιλήσω αναγκαστικά τώρα. Είναι το σπίτι της Ευρώπης, House of Europe, στο Βερολίνο. Έχουμε και τα παλιά κτίρια που θα τα ξανανοικιάσουν. 3.636 ε, τετραγωνικά, το 1 τρίτο έχει το Κοινοβούλιο, το άλλα 2 τρίτα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτι άλλο που οδήγησε σε κάποιες συζητήσεις και το λέω έτσι με μια πρεπίθηση πραγματικά. Αν θέλουμε να μας παίρνουν σοβαρά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα πρέπει να έχουμε περσινά ξινά φυλάδια ε, ξεθοριασμένα και ξεπερασμένα. Θα πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σωστή ενημέρωση. 317 ε, τετραγωνικά επιπλέον θα νοικιάσουμε ε, για να δείχνουμε κάποιες ταινίε και να χρησιμοποιούμε και τα νέα μίντια για να ενημερώνουμε. Ένα εκατομμύριο ε, είναι ε, το νίκη 420 ευρώ ένα τετραγωνικό. Η γειτονιά εκεί το κέντρο του Βερολίνου που λέγεται Berlin Mitte είναι επίσης πανάκριβη. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επομιστεί το κόστος του 1 τρίτου 32,8 και το υπόλοιπο 67,2 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 100 και ε, περίπου 800.000 ουσιαστικά θα είναι το κόστος για το κοινοβούλιο, αλλά ο ιδιοκτήτης επενδύει 2,8 εκατομμύρια ευρώ στην υποδομή του κτηρίου για εξοικονόμηση ενέργειας, ε, ανακαίνιση διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων, πράγμα που στο ειδινικές θα μειώσει το ετήσιο κόστος για μας. Οπότε θα πρότεινα να υποστηρίξουμε και αυτό το έργο. Or... Συστήνατε λοιπόν να υπάρξει γνωμοδότηση ή απλώ μια έγκριση με ψηφοφορία εδώ. Όχι, γνωμοδότηση. Είστε υπέρ του να μην υπάρχει γνωμοδότηση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελευταίο λοιπόν κοινό, κέντρο έρευνας. Yeah. Ναι. Είναι πάντα ένα χαρμόσυνο κεφάλαιο αυτό, γιατί είναι από τα πιο αποτελεσματικά όργανα μας και στα κτηριακά. Βέβαια, το κτίριο και το οικόπεδο είναι αρκετά ευαίσθητο και έχουμε τώρα νέες ρυθμίσεις και προδιαγραφές ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος της εισόδου προσωπικού ή ε, της προμήθειας αγαθών ε, σε χώρους που έχουν πυρηνικές ε, καταστάσεις. Και μέχρι τώρα ο έλεγχος που γινόταν στα πρόσωπα και στα υλικά ήταν ο ίδιος πάνω κάτω. Αυτό πλέον απαγορεύεται. Ε, θα έχουμε δύο ξεχωριστά κτίρια τώρα, αλλά επειδή είναι στην κατάσταση που είναι τα παλιά κτίρια, είναι επίγουσα η κατάσταση, είναι πραγματικά φρικτή εικόνα τα ίδια και μόνη μου η διεισόμαση τα κτίρια αυτά, οπότε... Εκεί που περνάει το προσωπικό και ε, οι επισκέπτες θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ε, είσοδος και χωριστό ε, κτίριο για ε, τα εμπορεύματα που εισάγονται. Θα πρέπει να είναι αυξημένη ασφάλεια. Θα πρέπει να ξεχωριστούν τα υλικά που είναι και ραδιενεργά από το προσωπικό και τους ε, επισκέπτες. 3,265 εκατομμύρια είναι το κόστος και επίσης 2,37 780.000 ευρώ για τα τεχνικά και τις συμβουλές 1,6 εκατομμύρια για τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ασφαλείας. Το συνολικό κόστος για το έργο είναι 5,6 εκατομμύρια επιπλέον του συνολικού κόστους. Υπάρχει και ένα αποθεματικό για έκτακτες δαπάνες 326.000 ε, ή 27 δεν θυμάμαι ακριβώς και η χρηματοδότηση θα προέρθει από ιδίους πόρους ε, του Ινστιτούτου και από την Ελβετία που συμμετέχει στο πρόγραμμα Ευρατών. Και μας έχουν στείλει τα στοιχεία εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχουμε νεότερα από πλευρά τους. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε Μόνικα. Δεν ξεκάθαρα. Υπάρχει κάποιο θέμα με αυτό. Ωραία. Η Επιτροπή ενημερώθηκε. Αυτό είναι το τέλος των ψηφοφοριών. Πάμε στα τελευταία δύο σημεία της σημερινής διάταξης. Πρώτα απ' όλα το 6, σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού αριθμός 1. Εδώ και 12 δεν είχαμε, εβδομάδες δεν είχαμε καμία, κανένα διορθωτικό προπολογισμό. Κυρία Γιάννη, αν θέλετε το λόγο. What point was it? Ε, Ah, Item 6 on the agenda. Σημείο 6 της διάταξης. Το σχέδιο διευθυντικού προπολογισμού είναι μια απλή υπόθεση. Αποτελεί τη συνέχεια της συμφωνίας για τα προγράμματα έρευνας και απλώς προβλέπει κονδύλια στις γραμμές του προπολογισμού τα οποία είναι μέρος της συμφωνίας. Έχουμε όμως μια τροπολογία από την Επιτροπή Βιομηχανία, διότι μία από τις γραμμές του προπολογισμού που συμφωνήθηκαν δεν ε, προκοδοτήθηκε με κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε η Επιτροπή Βιομηχανία αποφάσισε να υποβάλει αυτήν την τροπολογία για να βεβαιωθεί, να διασφαλίσει ότι υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση για αυτό το μέρος του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί. Απλώς το θέμα είναι ότι την τροπολογία αυτή θα πρέπει να τη συζητήσουμε σε τριμερή διάλογο, συγκεκριμένα στις 2 Απριλίου, και να αναβληθεί η ψηφοφορία για το σχέδιο διορθωτικού μέχρι τις 10 Απριλίου. Αφού συζητήσουμε και με το Συμβούλιο θα ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι μπορούμε να στηρίξουμε το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει διαφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Απλώς είμαστε βέβαιοι ότι, θέλουμε, ότι θα υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση, πλήρη χρηματοδότηση για όλα τα προγράμματα, ώστε να προχωρήσουν όπως προβλέπετε. Ναι. Επ' ευκαιρία ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν έχει τα στοιχεία τώρα στη διάθεσή της, γιατί μετά τη συμφωνία που πετύχαμε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει όχι με 170 πλέον, αλλά με 178 εκατομμύρια στη διεύρυνση του Ταμείου. Άρα το 2014 το ποσό θα ήταν λίγο υψηλότερο από εκείνο που είχε προβλεφθεί αρχικά. Νομίζω είναι 2 εκατομμύρια περισσότερα. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αλλάξει κάπως την πρόταση στο σχέδιο διαστατικού προϋπολογισμού ή θα το δείτε μόνο στον τριμερή διάλογο. Γιατί εκεί είναι 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ διαφορά που μπορεί να λυθεί βέβαια, αλλά δεν ξέρω πώς πρέπει να γίνει αυτό με διορθωτικό και συμπληρωματικό προϋπολογισμό, με τροποποίηση αυτού στον τριμερή διάλογο, ερωτώ. Okay, Θέλετε Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσετε στην ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τα δύο ζητήματα που τέθηκαν για το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 1 και την αλλαγή υπάρχει αλλαγή βάση και των όσων προβλέπονται για το 2020 για να αντικατοπτρίζει την νομική βάση και όπως μόλις αναφέρατε, υπάρχουν και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης έξω και θα υπάρχει και αύξηση στο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου. Πρώτα απ' όλα, βάση του Horizon 2020, του ιδιωτικού προπολογισμού, απλώς καλύπτει στον προπολογισμό του 2014 αυτή τη συμφωνία. Νέα κονδύλια μεταφέρονται σε αυτή τη φάση, ώστε να μην, υπάρξουν, να μην γίνει αμφιλεγόμενο το θέμα. Όμως με τη νέα δομή, όπω προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να μεταφέρει τα απαραίτητα κονδύλια, κυρίως με εσωτερικέ μεταφορέ, οπότε δεν υπάρχει καμία διαφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο προ το ποσό που θα μεταφερθεί. Απλώς εδώ ε, θέλουμε να βεβαιωθούμε. Καμιά φορά όμως το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Θέλουμε να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία εντός αυτής της θητείας του Κοινοβουλίου, δηλαδή με την Ολομέλεια του Απριλίου. Εάν γίνουν αλλαγές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να προλάβουμε να συμφωνήσουμε για να συμφωνηθούν και οι τροπολογίες που θα υποβληθούν και να περάσει και από την έγκριση της Ολομέλειας τον Απρίλιο η συμφωνία. Το ίδιο Ισχύει και την αύξηση στο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να αλλάξει την πρότασή τη. Αλήθεια είναι ότι το ποσό αφορά τα μερίσματα που ακόμα ε, πρέπει λοιπόν να φτάσουμε στο ποσό που αρχικά είχε οριστεί. Απλώς θα δούμε στο τέλος αν χρειάζεται να επανέλθουμε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι να αλλάξει το ιδιωτικό προπολογισμό, δομή υπάρχει, διάρθρωση υπάρχει για τον προπολογισμό, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού υπάρχει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, απλώς σε αυτή τη φάση θα δούμε εάν γίνεται μέχρι το τέλος του χρόνου, χρειαστούν πόροι και αν είναι διαθέσιμοι τέτοιοι πόροι αναδίπλωσης, θα κοιτάξουμε πριν το τέλος της χρονιάς να πάρουμε τις δεσμεύσεις, τις υποχρεώσεις τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για να γίνει προσαρμογή στη σωστή τετραετία, στην επόμενη τετραετία. Εκεί που πρέπει να γίνει δηλαδή άξιο του κεφαλαίου στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Το μήνυμα είναι να το έχουμε κατά νου και να μην ξεχνάμε το χρονοδιάγραμμα ώστε οι τροπολογίες για το 2014 να ισχύσουν. Ευχαριστούμε. Σας ικανοποιεί αυτό κύριε Συγγήτρια. Θα προσπαθήσω, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχει ολοκληρωθεί αυτό πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να το δούμε σε τριμερή διάλογο. Δεν μπορεί να συζητηθεί στις 25 Μαρτίου. Αλλά στις 2 Απριλίου, θα, αν προλάβουμε, θα μπορούμε στις 10 Απριλίου να ψηφίσουμε. Όπως υπόθηκε, δεν είναι ζήτημα ουσίας. Απλώς πρέπει να βρούμε τον σωστό τρόπο. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και με το σημείο 6 και το τελικό σημείο στην εμείς διάταξη είναι το σημείο 5, έγγραφο εργασίας για τα πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις στο πλαίσιο του υπολογισμού 2014 και 2015. Και πάλι η Ίντα και η κυρία Γιάννησεν είναι οι συγκεκριές. Ποια θέλει να ξεκινήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζετε ότι είναι παράδοση εδώ να έχουμε ένα έγγραφο εργασίας για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Ε, είναι μια παράδοση των τελευταίων ετών να πούμε ποια σημασία έχουν αυτά, ποιοι είναι οι στόχοι ε, που θέλουμε να επιτύχουμε και να καλύψουμε με αυτές τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου και ένα ε, χρονοδιάγραμμα ειδικό αυτή τη φορά γιατί έχουμε την ε, διακοπή των ευρωεκλογών. Είναι μικρή η προθεσμία, πιέζει βέβαια για να μπορέσουν οι παλιοί βουλευτές πριν φύγουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και μετά οι καινούργοι που παρόλο που είναι πολύ φρέσκοι να έχουν ένα δεκαήμερο για να κάνουν τις προτάσεις τους. Σε αυτό το έγγραφο εργασίας επίσης συμπεριλαμβάνεται μια πρώτη έκθεση ε, διάμεση βέβαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που εγκρίθηκαν για τον προϋπολογισμό του 2014. Αυτό είναι περισσότερο αμμοδιότητα της κυρίας Γένσεν, να το εξηγήσει εκείνη, θα το αφήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά είναι το σύνηθες κλασικό έγγραφο που έχουμε κάθε χρόνο για να εξηγούμε αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστούμε, Ιντε. Αν... Νομίζω όλοι δεχτήκαμε κρούσεις από όσους ενδιαφέρονται ιδιαίτερως φέτος για αυτό το θέμα, για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Νομίζω ο κατάλογος των πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων βάσει της συνηθισμένη διαδικασίας τα κανονικά έτη, είναι πολύ ωφέλιμη, διότι είδαμε ότι από τα 66 προγράμματα, 60 είναι στην σωστή στις σωστές διαστάσεις έχουν υπολογιστεί σωστά. Δεν ε, χρειάζονται λοιπόν οι παλιοί αγώνες που έπρεπε να δώσουμε. Διότι εντωμεταξύ υπήρξε χρόνος ώστε και, με, και οι συναδελφοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Βέβαια κάποιες φορές αυτό που συνέβη είναι ότι μια καλή ιδέα ήδη καλύπτεται από μια νομική βάση. Και αυτό ήταν και το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς κάποια από τα πιλωτικά προγράμματα. Ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν ως πιλωτικά προγράμματα γιατί τα κονδύλια θα μπορούσαν να φύγουν από τη γραμμή για τα πιλωτικά προγράμματα προς τη γραμμή με τη νομική βάση. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το τροχαίο υλικό λόγου χάρη και την ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα. Αυτό καλύπτεται από τον τομέα της καινοτομίας και την ε, μεταφορά, και την πρωτοβουλία για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Shift αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα. Και υπάρχουν και άλλα προγράμματα που φαίνεται ότι θα πρέπει να περάσουν από το πλαίσιο των πιλωτικών προγραμμάτων κάπου αλλού. Από το πλαίσιο δηλαδή πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων. Αυτό συμφωνεί με όσα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ψηφίσουμε τον προπολογισμό. Κάποιες φορές λέμε ότι είμαστε δημοσιονομική αρχή και αποφασίζουμε εμείς, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλό είναι να το θυμόμαστε. Ε, εάν κάποιοι συνάδελφοι είναι υποκινητές ε, των προγραμμάτων αυτών, καλό θα ήταν να έρθουν σε επαφή με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση και να το δουν το θέμα. Να είναι βέβαιοι για το τι συμβαίνει και να κοιτάξουν κατά πόσον όλα πηγαίνουν καλά και εφαρμόζονται. Πάντως η συνήθις διαδικασία έχει δείξει ότι δίνει καλά αποτελέσματα. βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί η υλοποίηση των πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων και ότι είναι πραγματικά νέε καινοτόμε ιδέε που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν αλλιώ από τον προπολογισμό ή από δυσονομικές γραμμές που έχουν νομική βάση. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κάποια πειθαρχία φέτο γιατί το προηγούμενο κοινοβούλιο μπορεί να προλάβει να δώσει κάποιες ιδέες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προλάβει να τις εξετάσει. Πάντως πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς θα κάνουμε, το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι νέοι συνάδελφοι ίσως να ενημερωθούν για τις ιδέες τους και να έχουν μια γρήγορη ενημέρωση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Διότι είναι πολύ δουλειά να κάτσει κανείς να επινοήσει και να σκεφτεί, να συλλάβει ένα πρόγραμμα και τελικά να μην γίνει τίποτα. Πάντως τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αυτά είχαν να πω Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αν έιντε. Κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει. Όχι, ας περάσουμε στα διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. Λίγη συνεδρίαση. <laughs>